Ε, για την ελευθερία του τύπου στην Κένια. Τον λόγο τον έχει ο κύριο Ματσάκη, σαν συντάκτη ε, του ψηφίσματο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η ελευθερία του τύπου ε, είναι ταυτόσιμη με την ελευθερία έκφραση. Αυτό βέβαια δεν εφαρμόζεται στην ιδανική, σε, ιδανικά σε, στην δική μας ε, κοινότητα, ε, διότι τώρα πολλοί ε, παραβιάζουν αυτή την ελευθερία ε, έκφραση οι διάφοροι βαρώνοι του τύπου, οι διάφορες πολιτικές αρχές και αυτό γίνεται και στις ΗΠΑ και σε κάποια κράτη της Ευρωπαϊκής Όνεσης. Αλλά όσον αφορά τουλάχιστον την νομοθεσία, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στις, κοινο, στις μας έχουν θεωρητικά την προστασία ουσία του νόμου για να λειτουργήσουν όσο οδοδόν πιο ελεύθερα. Και εδώ διαφέρουμε με την, με την κυβέρνηση, από την κυβέρνηση της Κένιας που εισάγει ε, κάποιες νομοθετικές ρυθμίσεις ε, έτσι ώστε να ε, μπορέσει να παρεμβαίνει και να καταδιώκει τα μέλη του τύπου. Γι' αυτό θα πρέπει να παρέμβουμε και να ζητήσουμε από την ε, κυβέρνηση της Κένιας να λειτουργήσουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με τον πιο δημοκρατικό τρόπο ε, και να αρθούν οι αυτές οι διατάξεις. Ελπίζουμε και εμπιστευόμαστε ότι η έκκληση που απευθύνουμε μέσω αυτού του ψηφίσματος θα αντιμετωπιστεί ε, όχι σαν μία παρέμβαση αλλά σαν μία φιλική συμβουλή που δίδεται προς την κυβέρνηση της ε, Κένιας και θα ληφθεί υπόψη από την κυβέρνηση αυτή και θα, η οποία θα επανεξετάσει όλα όσα έχει κάνει μέχρι τώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκέριγκερ Ντε Όντενμπεργκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Κένια περνάει μια σοβαρή πολιτική κρίση. Ο πρόεδρος Κιμπάκη ε, παραβιάζει την ελευθερία έκφραση και την ελευθερία του τύπου. Παραβιάζει τον Αφρικανικό, τον Αφρικανικό χάρτη ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δικαιωμάτων των λαών. Και πρόσφατα ε, έδωσε τη σύμφωνη γνώμη του για το τροποποιητικό νομοσχέδιο του 2008 σχετικά με τις επικοινωνίες ε, που οδηγεί και σε κατάργηση ε, σταθμών, τηλεοπτικών, ραδιοφωνικών κτλ. Η διεθνής κοινότητα θεωρεί ότι αυτό αποτελεί ένα μέτρο λογοκρισίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Παρά τις υποσχέσεις που έδωσε ο πρόεδρος, θεωρεί ε, ότι ε, ο πρόεδρος ε, ήρθε σε αντίθεση και με τον πρωθυπουργό της χώρας. Κάτι το οποίο θεωρούμε ότι δείχνει ότι η χώρα αυτή αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα. Εμείς θα πρέπει να ενισχύσουμε όλες ε, τις ε, δημοκρατικές ε, δυνάμεις στη χώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προωθήσει και να ενισχύσει όλες τις δημοκρατικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται στην χώρα. Ταυτόχρονα θα πρέπει και η κυβέρνηση της Κένιας να καταβάλει ε, δυνατή κάθε δυνατή προσπάθεια για να επανέλθει στο... σε μια φυσιολογική κατάσταση η... η χώρα. Με τον τρόπο αυτό πιστεύουμε ότι θα μπορούσε να σταθεροποιηθεί η κατάσταση στην χώρα και να αποφευθεί και η ανθρωπιστική καταστροφή. Ο κύριος Μπούρκε. Διάβασα αυτό το τροποποιητικό νομοσχέδιο το οποίο προσυπέγραψε ο πρόεδρος ε, Κιμπάκη. Έρχεται σε πλήρη αντίθεση και με, την Αφρικα, με τον Αφρικανικό Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δικαιωμάτων των Λαών και με οποιαδήποτε ε, διακήρυξη ή κείμενο προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πιστεύω ότι το, το κείμενο αυτό, το νομοσχέδιο αυτό ε, θα επιτρέψει την κατάργηση και το κλείσιμο ε, τηλεοπτικών σταθμών, ραδιοφωνικών σταθμών, εφημερίδων. Ε, ο πρόεδρος Κιμπάκη θα πρέπει να ακούσει την, την έκκλησή μας και να αποσύρει αν θέλετε αυτό το νομοσχέδιο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τι σημαίνει η ελευθερία του τύπου. Είναι ελευθερία της, εκ, της έκφρασης. Θα πρέπει να γίνουν προσπάθειες έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια κάποια συνένεση στην χώρα αυτή, να δημιουργηθούν ελεύθερα, μέτρα, ελεύθερα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να μην υπάρχει παρέμβαση στο έργο των μέσων αυτών. Επίσης θα πρέπει αυτοί οι οποίοι ε, οδήγησαν σε, στην βία της χώρα, την χώρα αυτή μετά τις εκλογές να ε, προσαχθούν στην δικαιοσύνη. Θα πρέπει να γίνουν περαιτέρω έρευνες, ανακρίσεις, διότι τον Δεκέμβρη του 2007 είδαμε τι είχε γίνει. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Μάιερ η, είναι πάρα πολύ βίαιη η ιστορία της χώρας για το δεύτερο παγκοσμίο πόλεμο σιγά σιγά δέχτηκαν οι Ευρωπαίοι ότι θα πρέπει οι Αφρικανικές χώρες σιγά σιγά να ανεξαρτοποιηθούν η Κένια όμως ήταν όπως και η Ζιμπάμπουε εξαίρεση οι επικοιοκράτες θεώρησαν ότι είναι πολύ σημαντικά τα οικονομικά τους συμφέροντα ούτως ώστε να τα αφήσουν στα χέρια των μαύρων όλα αυτά τα πλούτη. Πάντως υπήρξε μια αντιπαράθεση, ένα αιματοκύρισμα. Είχαμε το κίνημα απελευθέρωση των Μάο Μάο και εκεί βρίσκονται οι ρίζες των σημερινών ταραχών και συγκρούσεων. Είχαμε εκλογική νοθεία και παρά το ότι ε, μία παράταξη κέρδισε τις ε, εκλογές δεν την άφησαν να κυβερνήσει. Πάντως υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ και αντίθετα με τη Ζιμπάμπου ας θεωρήσουμε ότι στην Κένια υπάρχει περιθώριο συμβασμού κάποτε θεωρήθηκε σαν παράδειγμα προς στην Αφρική. Άνθιζε η επιχειρηματικότητα, υπήρχε σχετική ευημερία, όμως τώρα έχουμε καταστολή, φήμωση του τύπου, οικονομικά προβλήματα και Ήδη τώρα υπάρχει ε, οικονομική ασφυξία, υπάρχουν, ε, έχει επιβληθεί απαγόρευση κυριότητας πάνω από 40.000 τετραγωνικά μέτρα. Εν πάση τώρα θα πρέπει η αυταρχικότητα του Πρωθυπουργού να συγκρατηθεί. Άρα θα πρέπει να ε, περάσει το ψήφισμα και να υπάρξει κάποια εκλογική κατάσταση. Έχετε το λόγο για ένα λεπτό, κύριε Τάνοκ. Κύριε Πρόεδρε, η Κένια είχε τη φήμη ε, χώρας δημοκρατικής ε, με ελευθερία του τύπου. Ο πρόεδρος Κιμπάκη θα πρέπει να καταλάβει ότι ε, οι διάφορες ελευθερίες ενισχύουν η μία την άλλη και αυτό το οποίο προτείνεται τώρα δεν ταιριάζει σε έναν υπεύθυνο χώρας που ήρθε στην εξουσία διακηρύσσοντας τις αρχές της δημοκρατίας. Δυστυχώ, φαίνεται ότι δεν είναι ακόμη σε θέση να τηρήσουν τι αρχέ του ελεύθερου τύπου και τη Δημοκρατία. Ελπίζω ο πρόεδρος Κιμπάκη να ακούσει τι συμβουλέ μα και να αλλάξει άποψη. Αυτό θα μα καθησυχάσει σχετικά με την πρόθεση τη Κένια να δώσει την εξουσία σε μια ε, αρχή στην διακυβέρνηση, ούτω ώστε να έχουμε μια ευρύτερα ασφαλή περιοχή. Ε, χαιρετίζουμε την ε, ανακοίνωση του Προέδρου ότι θα κάνει διαβουλεύσεις με τα μέσα ενημέρωση και θα δώσει περισσότερε ελευθερίε. Ο ε, κ. Σοντίνγκα και το κόμμα του είναι κατά αυτού του νομοθετικού μέτρου και ε, θα πρέπει να ε, μην επέλθουν περαιτέρω διαιρέσεις στη χώρα λόγω της διαφοράς μεταξύ των κομμάτων. Η κυρία Στήλε, δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι που μου δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσω για αυτό το κοινό ψήφισμα για την ελευθερία του τύπου στην Κένια. Πριν από ένα χρόνο, όπω και άλλοι, και εγώ είχα απογοητευτεί, διότι μετά από τι αποτυχημένε εκλογέ στην Κένια, μετά από εθνοτικέ καθαρίσει και πολλέ διαδηλώσει, με θύματα πάνω από χίλια άτομα και ενώ έμειναν άστεγοι πάνω από 3.000 άτομα, ε, ξέρουμε ότι θα πρέπει να προσαφούν ε, οι υπεύθυνοι αυτών ε, που έγιναν πέρυσι και να γίνουν προσπάθειες να επανέλθει η δημοκρατία στην Κένια. Σε αυτό το πλαίσιο είναι πολύ αρνητικό το ότι στις 2 Ιανουαρίου ο πρόεδρος Κιμπάκη υπέγραψε το νομοσχέδιο για την τροποποίηση του νόμου του 1998 σε σχέση με τα δικαιώματα, με την ελευθερία του τύπου, γιατί με το τωρινό νομοσχέδιο υπάρχουν δύο τμήματα που επιβάλλουν λογοκρισία, άμεση λογοκρισία από την κυβέρνηση. Το τμήμα 88 δίνει στην κυβέρνηση σημαντικές δυνάμεις να διαλύει κανάλια ή ραδιοτηλεπτικούς σταθμούς που θεωρούνται ε, απειλή προς το κράτος και το τμήμα 46 δίνει τη δυνατότητα στο κράτος να διακόπτει εκπομπές οι οποίες μεταδίδονται από τα μέσα ενημέρωσης και οι δημοσιογράφοι και ο Πρωθυπουργός Οντίνγκα και από το κόμμα ODM ε, αντιτίθεται σε, αυτή, ε, σε αυτό το νομοσχέδιο είναι ατυχή η ψήφιση αυτού νομοσχεδίου και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες ε, οι διαφορετικές απόψεις που έχουν ακουστεί σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό η κυρία Πρόεδρε. Ήμουν μέλος της αλληλεγγύης στην Πολωνία και ξέρω ότι η ελευθερία του λόγου είναι η ανάσα της δημοκρατίας. Η κυβέρνηση της Κένια έχει υπογράψει και την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων Ανθρώπου και τα άλλα διεθνή κύματα για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου που περιλαμβάνουν και την ελευθερία του λόγου. Καταλαβαίνουμε τώρα ότι η Δυτικοαφρικανική Ένωση Δημοσιογράφων περιμένει να αλλάξει η απόφαση που συζητούμε. Και αυτό το ελπίζουμε και εμείς. Ελπίζουμε ότι η νομοθεσία για τα μέσα ενημέρωσης δεν θα αλλάξει έτσι ώστε να παραβιάζεται η αρχή της ελευθερίας του λόγου. Ζητώ από τις αρχές της Κένια να αλλάξουν την απόφαση σχετικά με την εισαγωγή ε, λογοκρισία στα μέσα ενημέρωσης και να σέβεται τα, τα δικαιώματα των μειονοτήτων και εθνικών και θρησκευτικών. Θυμόμαστε τι είχε γίνει πέρσι ε, μετά τις εκλογές στην Κένια όπου πάνω από 3.000, ε, όπου εκατοντάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και χιλιάδες διώχθηκαν από τις ε, από, την, από τα σπίτια τους. Ελπίζουμε όλοι οι υπεύθυνοι να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Έχω την κυρία Ζεύσκα, τον κύριο Ζεύσκα ως εκπρόσωπο σαν προσωπική αγόρευση. Κυρίε και κύριοι, είναι γεγονός ότι όντως κάποια ιδιωτικά μέσα ενημέρωση στην Κένια μετέσχον στην διάδοση αυτών των αρνητικών συναισθημάτων τούτο τόσο δεν είναι λόγος ε, να αρχίζουμε να επιβάλλουμε λογοκρισία διότι η ελευθερία του λόγου είναι το θεμέλιο της δημοκρατίας Η κατάσταση επιδεινώνεται από το γεγονός ότι στην Κένια το σύστημα των μέσων ενημέρωσης ήταν από τα καλύτερα στην Αφρική και αυτό δείχνει και αυτό, ε, δια, αυτό διαλύεται αυτή τη στιγμή. Κάτι που αντιβαίνει στην ελευθερία του λόγου. Η απόφαση παριθμών 36 μόνο αρνητικά μπορεί να λειτουργήσει. Ευχαριστώ. Συνάδελφοι, τώρα, γιατί μας ενδιαφέρει η ελευθερία του τύπου στην Κένια, γιατί συζητάμε το ζήτημα αυτό στα κατεπήγοντα ως παραβίαση των δικαιωμάτων ανθρώπου. Πρώτον, διότι η ελευθερία του τύπου είναι ένα βασικό ανθρώπινο δικαίωμα. Το λέει και η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, άρθρο 19. Η Κένια έχει υπογράψει την ε, ε, διακήρυξη αυτή και γι' αυτό πρέπει να σεβαστεί και το πνεύμα και το γράμμα. Πριν από ένα χρόνο, μετά τις προεκδικές εκλογές, οι διαδηλώσεις που μετατράπηκαν σε διεθνωτικές συγκρούσεις οδήγησε σε ε, πολλούς θανάτους και διωγμούς πολιτών και φιλών. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι η κυβέρνηση της Κένια και η Βουλή πρέπει να, αναδράσουν να δράσουν από κοινού σεβόμενοι την ελευθερία του τύπου και την ελευθερία του λόγου αλλά ταυτόχρονα τιμωρώντας και την ε, ατιμορρυσία και οδηγώντας του υπεύθυνους στο δικαστήριο. Κύριος Ματσάκης έχει το λόγο. Ενώ συζητάμε ανθρωπιστικά ζητήματα και ελευθερία τύπου σε τρίτες χώρες, να σας ενημερώσω πως ε, σύμφωνα με με ανταποκρίσεις από τη Γάζα τα γραφεία του ΟΗΕ που νωρίτερα σήμερα φλέγονται και όλη η βοήθεια η ανθρωπιστική που έχει στείλει αρκετή από αυτήν την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταστραφεί εντελώ. Το ίδιο ισχύει και για τα γραφεία του Reuters και ε, άλλων διεθνών πρακτορείων. Και συμφωνώ με την άποψη του Γενικού Γραμματέα, του κυρίου Μπαν Κίμουν, που είναι αυτή τη στιγμή στο Ισραήλ, ο οποίος είναι έξω φρενών από ό,τι λέγεται με τις Ισραηλινές αρχές. Ευχαριστώ. Κανονικά δεν θα έπρεπε να αποδεχτώ την παρέμβασή σα, κύριε Ματσάκη γιατί ο κανονισμό λέει πω όταν ζητάτε το λόγο με αυτή τη διαδικασία πρέπει να είστε επί του θέματο, από το οποίο ήταν η ελευθερία του τύπου στην Κέννη αλλά εν πάση περιπτώσει λόγω του ότι έτσι είναι η τραυματική κατάσταση το αποδέχομαι. Κύριε Αρέκτοβα, ο κύριος ένα λεπτό. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το ψήφισμά μας για την ελευθερία του τύπου στην Κένια εμφανίζεται σε μια πολύ ενδεδειγμένη στιγμή. Μιλούμε για δικαιώματα του ανθρώπου και για το τι συμβαίνει όταν αυτά καταστέλλονται από τη δικτατορία. Αυτό έχει σημασία για μας παρότι είναι εθνικό ζήτημα. Πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός ο Ντίνκα και ο πρόεδρος Κιμπάκη πρέπει να αναλάβουν δράση είναι εις βάρος της δημοκρατίας και δεν τον χρειάζεται η χώρα. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Κύριος Λίσκεβιτς. Κύριε Πρόεδρε, επί κομμουνισμού στην Πολωνία και σε άλλες χώρες υπήρχε ένας νόμος που έλεγε ότι οποιοδήποτε διαδίδει πληροφορίες που μπορούν να διαταράξουν τη δημόσια τάξη τιμωρείται. Ε, τέτοιες διατάξεις ήταν πολύ χρήσιμες ε, για τις αρχές και αυτό ήταν μάστιγα και για τον τύπο και για τους ιδιώτες, για τα άτομα. Βλέπουμε τώρα πως έχουμε παρόμοιες κινήσεις από πλευράς ε, Κένιας και δεν μπορεί να δικαιολογηθεί αυτή η λογοκρισία. Και αυτό το επιχείρημα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί λέγοντας πως πρέπει να φημωθεί ο τύπος γιατί θα διαταράξει την ειρήνη της χώρας. Γιατί η ελευθερία του τύπου είναι θεμελιώδης για τη δημοκρατία. Έχουμε τον Επίτροπο κ. Σπίτλο που θα απαντήσει εξ ονόματος της Επιτροπής. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θέλω Ευθύ εξ αρχή να υπογραμμίσω ότι η ελευθερία του λόγου συμπεριλαμβανομένων και τη τηλεόραση και του τύπου αποτελεί ένα από τους στυλοβάτες της ελευθερίας. Αποτελεί μια βασική ελευθερία στην Ευρώπη και δεν θα πρέπει να αμφισβητείται. Η πράξη επικοινωνία, ο νόμος για την επικοινωνία το 2008 που την 1η πρώτου 2009 έγινε ε, νόμος της Κένια περιλαμβάνει κάποια στοιχεία που πιθανώς παρα, ε, παραβιάζουν την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και γι' αυτό μας ικανοποιεί η πρόσφατη απόφαση του Πρόεδρου Κιμπάκη στις 2 Ιανουαρίου να αναθεωρήσει κάποια αμφιλεγόμενα μέρη αυτού του νόμου. Χαιρόμαστε που ζήτησε από τον Πρόεδρο, από τον Υπουργό Επικοινωνίας και τον Γενικό Εισαγγελέα να συναντηθούν με τους εκπροσώπους του τύπου για να συζητήσουν τροποποίησεις του νόμου αυτού που μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ανησυχίες. Η ελευθερία του λόγου και η ελευθερία του τύπου ανήκουν ε, ε, στην δημόσια, στο χώρο της δημόσιας διακυβέρνησης υπό την ευρία έννοια που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σαφώς πιστεύω ότι ο ελεύθερος και υπεύθυνο τύπος αποτελεί στοιχείο δημοκρατίας και της ενόμου τάξεως που βεβαίως αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της βιώσιμης ανάπτυξης. Ο διάλογος είναι ο τρόπος με τον οποίο ε, ο τύπος και η κυβέρνηση της Κένιας μπορούν να ε, να ε, συζητήσουν αυτό το θέμα. Πρέπει να εμπλακούν όλες οι ενδιαφερόμενες πλευρές και θα πρέπει τα μέρη να καταλήξουν σε συμφωνία και να βρουν τις απαραίτητες προτάσεις ώστε να τροποποιηθεί ο νόμος αυτός. Όσον αφορά τώρα την μετεκλογική βία, η Κομισιόν ε, χαιρετίζει την έκθεση της ε, Ανακριτικής Επιτροπής η οποία ζητά να εφαρμοστούν οι προτάσεις της έκθεσης μεταξύ των οποίων είναι και η σύσταση ενός δικαστηρίου στο οποίο θα έρθουν όλοι οι υπεύθυνοι για αυτή τη βία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπη και τώρα περνάμε αμέσως στη ψηφοφορία. Σύμφωνα με την ε, ημερήσια διάταξη θα ψηφίσουμε το, την πρόταση ψηφίσματος για το Ιράν, υπόθεση Σιρήν Εμπαντή. Ε, τίθεται σε ψηφοφορία ένα κείμενο το οποίο ε, αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες προτάσεις. Περ, κατά, αποχές, εγκρίνεται με